Good morning, everyone. Καλημέρα σε όλου. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη. είναι η έγκριση της ημερήσια διάταξης με την εξαίρεση του θέματο πρέπει που η κυρία Περές είναι η ανεβλήθη. Θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, σας προτείνω να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις. Αντιπροσωπή Ευρωβουλευτών, εμού συμπεριλαμβανομένου, της Επιτροπής αυτής, με την κυρία Σάραμπο. Πήγαμε στην Ιρλανδία λοιπόν και ε, όπως ξέρετε ξεκινά, ε, την ε, επόμενη Προεδρία που ξεκινά τον Ιανουάριο κατά διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε η Ιρλανδική οικονομία και η επιτυχής εφαρμογή της, ε, του προγράμματος εφαρμογής της χώρας. Αυτά συζητήθηκαν εκτενώς για την προσωπία αναγνώρισε τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιρλανδία ε, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και σημείωσε ότι πολλοί από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ιρλανδίας, κυρίως το υψηλό επίπεδο εκπαίδευση του πληθυσμού, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Και το πώς θα ανακάμψει η Ιρλανδία και πώς θα επιλύσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την τραπεζική κρίση που πέρασε. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με προσωπικότητες της κυβέρνησης και πήγε και στο Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας, Κεντρική Τράπεζα, και εκπρόσωποι του χρηματοδοτικού τομέα στο Δουβλίνο συναντήθηκαν μαζί μα και διάφοροι γενικά ενδιαφερόμενοι φορεί συμμετείχαν συζητήσει. Ο Ιαν Χέστιτ, ο υπουργό Οικονομικών, μίλησε μαζί και ο κ. Κράιτον, ο υπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνομίλησε μαζί μας. Και τον κύριο Χόγκαν και τον κύριο Αντέλφε συναντήσαμε διοικητή και υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για να συζητήσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προβλήματα των χρηματοστατικών μεταρρυθμίσεων για να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Συζητήσαμε το θέμα διαπραγματεύσεων προτάσεων για να έχουμε ενιαία εποπτεία των τραπεζών και αύριο θα ψηφίσουμε τη σχετική έκθεση εδώ όπως γνωρίζετε. Άλλες ανακοινώσεις θα τις κάνει η κυρία Πρόεδρος το απόγευμα, στην απογευματινή συνεδρίαση. Πάμε αμέσως λοιπόν στο πρώτο σημείο της σημερινής διατάξεως, πρόταση οδηγία του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2006-112 ΕΟΚ όσον αφορά ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ ως μηχανισμός ταχείας αντίδρασης καταπολέμησης των απατών ΦΠΑ. Ο κ. Ντέιβιτ Κάζα είναι συγγητής. Εκ μέρου του κ. Κάσα θα μιλήσει ο κ. Γκοζέ. Κύριε Γκοζέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και 15 μέρε ήμουν η κυρία Λούλινγκ. Σήμερα είμαι ο κ. Κάζα. Βλέπετε ποικιλομορφία που μπορεί να εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Ντέιβιτ μου άφησε κάποιες σημειώσεις, να σας εξηγήσω ποια είναι η θέση του. Το κείμενο που προτείνεται από την Επιτροπή προορίζεται στο να καλύψει τα κενά του παρόντος συστήματος για την καταπολέμηση των απατών του ΦΠΑ και που βασίζεται στο μηχανισμό αυτορύθμισης που δεν ήταν αποτελεσματικός μηχανισμός. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μηχανισμού ταχείας αντίδρασης με στόχο την καταπολέμηση, την ταχεία καταπολέμηση της απάτης στον τομέα αυτό του φόρου θέμες αξίας και θα συμπληρώνει το σύστημα των παρεκκλήσεων που υπάρχει. Ο Ντέβιτ Κάσα υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές μέσω διαβουλεύσεων όμως με τους διαπίστωσε ότι κοστίζει ο μηχανισμός αυτό ε, παραγωγής ρευστού, χρήσης του ρευστού και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ ακραίες περιστάσεις αυτός ο μηχανισμός. Και η τροπολογία 6 αντικατοπτρίζει αυτό το θέμα. Θεωρεί ότι δεν είναι επίμαχο το θέμα αυτό της ίσως του συστήματος Γαϊτανάκη του ΦΠΑ για την απάτη ε, και οι προτάσεις ε, έγιναν, κάποιες προτάσεις έγιναν και αναμένονται από τους συναδέλφους για να βελτιωθεί το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν επιτρέπετε να σας πω και κάτι, μια ιστοριούλα. Μιλούσα την περασμένη φορά σαν κυρία Λούλινγκ, αλλά η έκθεση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν το ανέφερε και θεώρησε ότι εγώ έθεσα όλα τα ερωτήματα που είχε θέσει η κυρία Λούλινγκ. Οπότε ήρθε επίτροπος για να προσπαθήσει μαζί μου να κουβεντιάσει για να δει αν έχουμε διαφορέ. Εγώ του είπα ότι δεν έχω διαφορέ μαζί σα, αλλά ήταν η κυρία Λούλινγκ με το πνεύμα που τη χαρακτηρίζει και με τη λογική που ακολουθεί, που οδηγήθηκε σε διάφορε ερωτήσει και εγώ απλώ ήμουν πιστό φερέφων αυτή. Ο κ. Κάζα δεν έκανε εκ παρατηρήσεις, οπότε δεν θα ενοχλήσω ξανά τον Επίτροπο τον κύριο Σεμέτ όσον αφορά την φορολόγηση. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Ευχαριστούμε. Το ΕΛΚ είναι τυχερό να έχει έναν συντονιστή τόσο ευέλικτο όσο εσάς. Και εξ ονόματος των σοσιαλιστών θα λάβει τον λόγο. Λούτβιξον. Εξ ονόματος Λούτβιξον στην κυρία Φερέρα. Και πάλι η σοσιαλιστική ομάδα έχει την τύχη να έχει εσά ω συντονίστρια. Κυρία Φερέρα, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Παίρνω τον λόγο εξ ονόματο ε, του κυρίου Λουμπλιχία που δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Ω σημείο αφετηρίας και αυτή είναι η άποψη του Όλε, αυτή η σημαντική πρόταση θα πρέπει να ε, γίνει θερμά δεκτή η καταπολέμηση της, ε, κατα... της απάτης ε, και της διαφυγής είναι σημαντική υπόθεση. Πέρα από την πρόσθετη αξία, πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν σε αυτό το τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας ένα μηχανισμό άμεσης αντίδρασης. Είναι ένα σκόπιμο πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια λογική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιες φορές ε, τα κράτη-μέλη και δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να δράσουν αρκετά ταχαίως κατά της απάτης ΦΠΑ. Ο κύριος Λούτβιξον με χαρά βλέπει ότι ο κύριος Κάζα συμμερίζεται αυτές τις θετικές προτάσεις της έκθεσης και είναι πεισμένος ότι το κοινό έργο αμφωτέρων και των δύο για αυτό το θέμα στις επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ επικοδομητικό ζήτημα, θα προχωρήσει θετικά. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει ο Λε ότι υπάρχει εδώ ημιτελές έργο γύρω από αυτή την πρόταση και πρέπει να ολοκληρωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει καλύψει όλη την απόσταση. Πρόσθετα στοιχεία χρειάζονται, ιδιαίτερα γύρω από δύο κύριους άξονες. Πρώτο, πρώτος είναι ότι ο μηχανισμός ε, αναδρομικής ε, επιβάρυνσης είναι ο μόνος μηχανισμός καταπρέμψης απάτης σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το τέλος της διαδρομής. Δεν είναι αποδεκτό να μην υπάρχει ένα πιο εξειδικευμένο σχέδιο πώς θα προσθεθούν νέα εργαλεία στην εργαλειοθήκη αυτή τα επόμενα χρόνια στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει μια στερεά αξιολόγηση και δεσμεύσεις ώστε κλιμα... κλιμακωτά σταδιακά να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεύτερον, η πρόταση δεν είναι ιδιαίτερα επικοδομητική όσον αφορά την διασφάλιση συντονισμού μεταξύ κρατών μελών με την εφαρμογή ενός ειδικού μέτρου όπου θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις ένα κράτος μέλος στο ΦΠΑ άλλων κρατών μελών. Αυτό είναι κέρια σημασία θέμα όταν θέλουμε ο μηχανισμός αυτός να λειτουργήσει καλύτερα στην πραγματική ζωή, πιο αποτελεσματικά σε σύνδεση με αυτά τα οποία κάνουν τα κράτη-μέλη που έχει θεμελιώδη σημασία το θέμα. Ο Λελούνιξον θα ήθελε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλους, σε όλα τα βήματα και τις κλίμακες ε, για αυτούς, για αυτούς τους μηχανισμούς από τα κράτη-μέλη. Αν δει κανείς συνολικά σφαιρικά το τι διεξάγεται, η συνεργασία, η προσαρμογή, ο συντονισμός θα διευκόλυνε τα πράγματα. Επίσης, ο συνάδελφος θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει με συμπληρωματικές προτάσεις για αυτή την πτυχή μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο. Όσον αφορά τις προσπάθειες ε, του κ. Κάτρας, ποιες ε, προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η απάτη μέσω στατιστικών στοιχείων, ο κ. Όλε πιστεύει ότι αυτό πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά Κάποια πρόσθετη αποσαφήνιση θα μπορούσε να είναι θετική. Ο μηχανισμός της ταχεία αντίδρασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται, ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα κράτη-μέλη μπορούν προληπτικά να δράσουν για την καταπολέμηση απολειών ΦΠΑ στο άμεσο μέλλον όπως θα μπορούσε να αναμένεται και γι' αυτό στατιστικά θα πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να αναφέρεται. Ο Όλε πιστεύει τέλος ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε μια πιο ισχυρή διατύπωση για τους πόρους και τη διοικητική ικανότητα των αρχών ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης θα μπορέσει να λειτουργήσει ικανοποιητικά μόνο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση σε όλες τις χρονικές στιγμές άμεσα και αποτελεσματικά να λαμβάνει μέτρα και να δρά. Πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό και το υλικό να επαρκεί ώστε η διαδικασία λήψης απόφασης θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πράγματα αποτελεσματικά. Μετά από αυτά τα σχόλια του κ κυρίου Όλεγ επίσης θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον κύριο Κάζα για ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης και προσβλέπει και αδημονή να συνεργαστεί επ' αυτού του χαρτοφυλακίου μαζί του. Ευχαριστώ. Σε... Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φερέρα. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, η κυρία Κλέβα παρακαλώ. Όχι. Α, εντάξει. Συγγνώμη. Ε, δεν υπάρχει κανείς εξ ονόματος των φιλελευθέρων και σε σχέση με τον κύριο Γκίγκορτ δίνω τον λόγο εξ ονόματος της κυρίας Λι παρακαλώ έχετε τον λόγο Ευχαριστώ πολύ μιλάω για τον εαυτό μου θα χαίρεστε που τα ακούτε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάζα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή έχω δύο παρατηρήσεις αν επιτρέπετε πρώτον Συμφωνώ ότι βλέποντας τις ευρύτερες ε, συνέπειες του αναδρομικού τέλους για τις επιχειρήσεις και του συστήματος ΕΠΑ, ένας μηχανισμός ταχείας αντίθεσης που χρησιμοποιείται σαν τελευταίο ε, άμυνα όταν άλλα τα μέτρα καταπολέμησης των απατών μέσω των δυσίμων ε, μέσων έχουν αποτύχει. Τα κράτη δεν θα πρέπει να πηγαίνουν σε αναδρομικό τέλος και να, υποκαθιστά αυτό μια καλύτερη εξολόγηση κινδύνου. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω αφορά την τροπολογία 6. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερες συζητήσεις για το όσον αφορά την ξαφνική απάτη μεγάλης κλίμακας. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθοριστεί αυτό. Φοβάμαι μην ακολουθήσουμε τη διαδρομή που προτείνει ο εισηγητή που επιτρέπει αναδρομικό τέλος όταν περαστεί, ξεπεραστεί όριο απάτης. Εάν υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός, ε, χρειάζεται ευελιξία. Και αν τα κριτήρια είναι αυστηρά, θα γίνει άκαμπτος ο μηχανισμός. Ε, και δεν ξέρουμε αν είναι σωστό το ποσοστό που θα καθοριστεί. Περιορίζεται το περιθώριο λιγών των κρατών μελών που ίσω θα πρέπει να κινηθούν εκ των προτέρων πριν υπάρχουν σημαντικέ απώλειε για να σταματήσει το πρόβλημα έγκαιρα. Βασίζεται και επί στατιστικών στοιχείων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα μέχρι ότου περάσει το γεγονό. Και επειδή χρειάζονται και προσαρμογέ και τελικά να, συλλεχθούν και τα στατιστικά για το ΦΠΑ που έχει συλλεχθεί και αυτό οδηγεί σε επιβράδυνση ε, και ίσως τελικά να υπονομευθεί το μέτρο και τίποτα υπάρχουν και προσφυγές. Παρ' όλα αυτά η έκθεση είναι πολύ καλή και προσβλέπω σε συνεργασία με τον David και τους άλλους κοιόδης για την ολοκλήρωση του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Η κυρία Κλέμπερ έχει το λόγο. Yes, speaking on Ναι, μιλάω και εγώ εκ μέρους του εαυτού μου, μέλος του S&D είμαι. Θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ τον εισηγητή ε, που συνέταξε αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Ετοιμάζω μια γενικότερη έκθεση για φοροδιαφυγή και φορολογικές απάτες. Ε, θα υποβληθεί προς το τέλος του έτους αυτή. Αυτό είναι σε αντίδραση του σχεδίου δράσεως που υποσχέθηκε σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να πω μερικά πράγματα όσον αφορά το μηχανισμό ταχείας αντίδρασης κατά των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Σαν πρώτο βήμα στην καταπολέμηση των απατών που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη που προτείνει και ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι πρόσδεκτη και να υποστηριχθεί. Αλλά θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από συνάδελφοι λεπτομερέστερο σχέδιο δράση όσον αφορά την φοροδιαφυγή και τι φορολογικέ απάτε, κάτι που θα ξεπερνά το μηχανισμό αυτό τη ταχεία αντίδραση ακόμα και για την αντιμετώπιση των απατών ΦΠΑ αυτών καθεαυτών. Και όταν βλέπουμε τα βραχυπρόθεσμα εργαλεία που υπάρχουν, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από τον προτινόμενο μηχανισμό. Η Ευρώπη χάνει, και το επαναλαμβάνω αυτό, όποτε μπορώ, ένα τρει ευρώ σε ενδεχόμενα φορολογικά έσοδα κάθε χρόνο και Τέτοιε απώλειε δημοσίου εισοδήματο, τέτοια περίοδο μεγάλη οικονομική κρίσεω και ε, διαφόρων περικοπών στα κράτη-μέλη είναι κάτι απαράδεκτο. Υποστηρίζω ένθερμα την προσπάθεια κάνει και ο Σκάζα για να υποβάλει συγκεκριμένου ορισμού. είναι βασικό στοιχείο χαρακτηριστικό της έκθεσης και συμφωνώ ότι μπορεί να βοηθήσουν ορισμοί όσον αφορά το θέμα της, των φορολογικών απατών. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους ορισμούς και ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα θα ήταν να συμπεριλάβουμε αναμενόμενες απώλειες στον ορισμό των απατών και επαναλαμβάνω τέλος αυτό που υπόθηκε για τη διαφάνεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του μηχανισμού ταχείας αντιδράσεως είναι να αντιμετωπιστούν περίπλοκοι μηχανισμοί απατών που ξεπερνούν πολύ συχνά ένα κράτος μέλος και αυτό υπόθηκε σήμερα τουλάχιστον τρεις φορές Οπότε ο συντονισμός μεταξύ κρατών μελών καθώς και διαφανής επεξεργασία ετοιμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί και να το έχουμε σίγουρο, να είναι εγγυημένο πριν προχωρήσουμε. Ευχαριστώ εκ νέου τον κύριο Κάσα για την έκθεση και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά τη σύνταξη τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. <clears throat> Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω. Λέει ο κύριος Κλούτε. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραμπόνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξή του στην πρότασή μας. Δύο-τρεις παρατηρήσεις γύρω από τις τροπολογίες σας. Πρόκειται για μια πρώτη θα έλεγα αντίδραση ή πρόκειται για την αντίδρασή μας συγκεκριμένα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν πρόκειται για έναν τακτικό λειτουργικό μηχανισμό. Πρόκειται για την αντιμετώπιση άμεσα ορισμένων συγκεκριμένων ε, συμβάντων. Ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν με τα πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα, πέντε δις απώλεια μέσα σε λίγες εβδομάδες λόγω των απατών. Γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα. Και οι εμπλεκόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα από τις απάτες αυτές. Πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα τέλη είναι περιορισμένα και ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τώρα, τι είναι μια μαζική απάτη, ορισμός δηλαδή. Ο εισηγητής αποπειράται επί τη βάση ποσοστών εσόδων να ορίσει το τι είναι κάτι τέτοιο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, ε, να το κάνουμε, να το πετύχουμε. Αφήνουμε αυτή την ευελιξία στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα μας ζητήσουν την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού άμεσης αντίδρασης σε πολύ σημαντικές κατεπίγουσες περιπτώσεις και μόνον. Θα πρέπει επίσης να πάρουμε και προληπτικά μέτρα, όχι μόνο να διαπιστώνουμε την απάτη και να αντιδρούμε, αλλά να προλαμβάνουμε την απάτη στην συγκεκριμένη περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων. Τώρα, για το εάν μια προσωρινή εξαίρεση είναι κάτι το εφικτό. Εμείς πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες λύσεις μόνιμου τύπου, για τις αντιδράσεις των κρατών μελών και ο Επίτροπος και μετά θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα καταπολέμησης των απατών πριν από το τέλος του έτους με συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως, για την καταπολέμηση των απατών στο ΦΠΑ, αυτό εξαρτάται από την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δράσει σαν συντονιστής μόνο, η πρωταρχική ευθύνη θα έλεγα ανήκει στα κράτη-μέλη. Τίποτα άλλο πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ραμπονή. Κύριε Γκοζές θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω ότι από πλευρά του Νταβίντ Καζά Σημείωσα τις παρατηρήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι είναι συγκλίνουσες και επικοδομητικές και ο Νταβίντ θα ανταποκριθεί στην ανυπομονησία ορισμένων για την εκκίνηση των συζητήσεων για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα επιτρέψουν τη βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Να θυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η πέμπτη ε, Δεκεμβρίου 12η μεσημβρινή εξέταση των τροπολογιών θα γίνει την 21η Ιανουαρίου του επομένου έτους και η ψηφοφορία στις 22 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τώρα κανονικά προβλέπεται να γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2013. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης βελτιωμένη συνεργασία στον τομέα <clears throat> του ε, φόρου ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η κυρία Ποδηματάμος δεν είναι μαζί μας. Ούτε και η Σκιώδης δεν είναι εδώ. Minutes. So we will... Κοιτάξτε, θα διακόψουμε Σας περιμέναμε. Ήρθε η κυρία Πολύματα. Περιμένουμε ένα πεντάλεπτο, αν θέλετε, για να δώσουμε κάποιο χρόνο. Ένα λεπτό, μάλιστα. Συζητήσαμε ε, γρήγορα το προηγούμενο θέμα, οπότε έχει νόημα περιμένουμε λίγα λεπτά για να περιμένουμε να έρθουν οι για το επόμενο θέμα. Παρακαλώ, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ποδηματά, η συγγήτρια για το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας ε, σε σχέση με τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ποδηματά. Συζητάμε τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί στη σύσταση για να επιτραπεί η ενισχυμένη συνεργασία γύρω από το θέμα της δημιουργίας ε, του φόρου αυτού χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές διότι ήταν ε, επαρκώς επικοδομητική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το θέμα. Εξ αρχής είπαμε ότι εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην αξιολόγηση του αν οι νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανόνων της ενισχυμένης συνεργασίας εκπληρούνται και ε, θα αποφύγουμε να μπούμε σε μια συζήτηση επί της ουσίας της, αναθεωρημένης πρότασης. Θα ακολουθήσει η συζήτηση μετά από την πρόταση την οποία θα κάνει η Επιτροπή Γι' αυτό λοιπόν να ευχαριστήσω τους Κιώδης και όλους τους άλλους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. Λάβαμε 28 τροπολογίες συνολικά. Να σας ενημερώσω ότι εγώ έχω προτείνει τελικά δύο συμβιβαστικές, οι οποίες θα έλεγα συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες της ενισχυμένης συνεργασίας και όχι με την ουσία της για να μπορέσουμε έτσι να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στην παρούσα φάση. Η πρώτη συμβιβαστική υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει ότι ο φόρος αυτός θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του εφόσον εισαχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σφαιρικό επίπεδο. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες να υπάρξει μια συμφωνία σε γενικότερο παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα λέμε ότι οι χώρες οι οποίες προχωρούν στην εισαγωγή της επιβολής ε, του φόρου αυτού μετά από την εφαρμογή των κανόνων της ενισχυμένης συνεργασίας θα αποτελέσουν το σωστό παράδειγμα γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι μη συμμετέχουσες χώρες να μην ε, προσελκυστούν ε, όταν ε, φανεί ακριβώς ε, το όφελος για τις χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τον φόρο αυτό. Και αυτό θα είναι ένα παράδειγμα για να εφαρμοστεί ο φόρος αυτός παγκόσμια. Η δεύτερη τώρα συμβιβαστική την οποία καταθέτω ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπληρώσει την αρχική μελέτη επιπτώσεων εξετάζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αυτού φόρου σε ορισμένες χώρες, σε ένα μικρότερο αριθμό χωρών, έτσι ώστε να προταρμώσει την αναθεωρημένη πρότασή του ανάλογα, <clears throat> πρότασή της μάλλον ανάλογα. Νομίζω ότι έχω ενσωματώσει προς την κατεύθυνση αυτή τις τροπολογίες 3 της κυρίας Λούλινγκ, 5, 12, 13, Ματίας Κλούτε, και αυτό ισχύει και για τη διατύπωση της πρώτης συμβιβαστικής και ταυτόχρονα ε, ζητάμε την ε, συμπλήρωση της αρχικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες Λούλινγκ μεταξύ άλλων. Να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εργάζεται προς την κατεύθυνση της συμπλήρωσης της αρχικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της εφαρμογής του φόρου αυτού σε χώρες που συμμετέχουν στο σχήμα και σε χώρες που απέχουν. Να προσθέσω εδώ ότι μας κάνει εντύπωση το ότι οι μη συμμετέχουσες χώρες ανησυχούν για τις επιπτώσεις της εισαγωγής του φόρου αυτού από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Τώρα, για τις υπόλοιπες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί, κάποιες από αυτές επαναλαμβάνουν τις θέσεις τις οποίες έχει υιοθετήσει το Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Μάιο. Αυτό ισχύει για την τροπολογία 4 του Ίνεν 15 Ματίας και Κλούτε και οι δύο αυτές τροπολογίες ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση επί τη βάση της εκθέσεως που υιοθετήσαμε το Μάιο και πρέπει να υποστηριχθούν. Ε, δεν εκπλησόμεθα βέβαια από το ότι υπάρχουν τροπολογίες που απορρίπτουν την ενισχυμένη συνεργασία. Έχουν κατατεθεί κυρίως από τους Σουηδούς συναδέλφους Ερκμαρκ, Σμιτ Να επαναλάβω εδώ ότι αυτό με εκπλήσει λίγο. Κάποιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι οι αντιτιθέμενοι στην εφαρμογή του φόρου αυτού θα ανακουφίζονταν ε, από την ε, διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας εφόσον ήθελαν να είναι συμβατοί με τα επιχειρήματα τα οποία είχαν καταθέσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε ξεκινήσει στις αρχές του χρόνου ότι ο φόρος αυτός θα ωφελούσε και τις δικαιοδοσίες και χώρες που δεν καλύπτονται από το επίσημο έβρος του. Και τώρα εκπλήσει λοιπόν το ότι οι βουλευτές αυτοί εκπλήσονται και ανησυχούν για διαφορετικούς λόγους. Απορρίπτουν την ενισχυμένη συνεργασία γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι τόσο επιτυχής η εφαρμογή του κανόνα αυτού που θα επηρεάσει αρνητικά τις μη συμμετέχουσες χώρες. Τέλος, θα ήθελα όλος εγκαρδίως να ευχαριστήσω τους σκιώδεις για την επικοδομητική του στάση να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Λούλινγκ γιατί πράγματι ακολούθησε μια πολύ επικοδομητική γραμμή αν και είναι πάρα πολύ γνωστό ότι οι προσωπικές της απόψεις δεν ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά έδρασε στα πλαίσια των τροπολογιών που κατέθεσε ως εκπρόσωπος της πολιτικής της ομάδας του ΕΛΚ. Πρέπει λοιπόν να κλείσει αυτή η διαδικασία σύμφωνης γνώμης έτσι ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η πραγματική συζήτηση επί της ουσίας του φόρου αυτού μια συζήτηση η οποία θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την παρούσα. Ευχαριστώ κύριε Ποδηματά. Η κυρία Λούλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι κατόπιν της δικής μου, λόγω της δικής μου απουσίας και άλλων για λόγους επαγγελματικούς εδώ και δύο εβδομάδες χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες που αφορούν την πρόταση διευρυμένης συνεργασίας. Παρά την πίεση του χρόνου, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε δεόντως τα διακυβεύματα, διότι τελικά ε, υπερβολικός ενθουσιασμός μπορεί να θολώνει κάπως ε, τη σκέψη κάποιων. Θέλω να το είπα στον αγαπητό συντονιστή την περασμένη φορά, σκοπός της διαδικασίας δεν είναι να ξαναρχίσουμε μια συζήτηση όσον αφορά τα, τα υπέρ και τα κατά μια συμφωνίας για χρηματοπιστωτικό φόρο. Ε, υπευλήθησαν 28 τροπολογίες και αρκετοί συνάδελφοι δεν είχαν κατανοήσει ότι πρέπει να ακολουθείτε με κοινή προσέγγιση και δεν θα πρέπει να δίνεται κάποια δεοντολογική έκφραση άποψης στις ε, αιτιολογικές σκέψεις. Και δεν έχουν, σκέψει, δεν έχουν θέσει τέτοιου είδους κρίση σε αυτή την έκθεση. Αυτό που μετρά είναι να μπορούμε να αποτιμήσουμε τις συνέπειες μιας ενισχυμένης συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη λειτουργία της ενίας αγοράς, συνέπειες που υπάρχουν για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν και συνέπειες για εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξή. ότι και τα κράτη-μέλη που θα επιθυμούσαν να πόσχουν από τον μηχανισμό τελικά θα πρέπει να ασχοληθούμε το θέμα επανειλημμένα, είπε ο Σεμέτα, ότι η πρόταση που θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εδράζεται κυρίως επί της αρχικής προτάσεως του 2011. Όμως αυτή η θέσπιζε αρκετά, προσέγγισε εξοεδαφική για να μην υπάρχει τρόπος ε, παράβασης των διαφόρων χρηματοστηρικών διαδικασιών. Και αυτό είναι ένα μέτρο προσέγγιση που αφορά το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουμε να ξέρουμε ποια θα είναι η εμβέλεια του εξοδαφικού ε, χαρακτήρα των συναλλαγών. Δεν γνωρίζουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις και τις διαπραγματεύσεις θα είναι περίπλοκες οι συζητήσεις και οι εργασίες, αλλά δεν μπορούμε να διατηνόμεθα ότι μόνο τα κράτη-μέλη που θέλουν τη συνεργασία αυτή θα επηρεάζονται από το όλο σχήμα. Αυτό δεν αληθεύει. Εάν έχουμε το συνδικό ίδρυμα ενός κράτους μέλους εκτός της συνεργασίας αυτής, πραγματοποίησε μια συναλλαγή επί αξιών που προέρχονται από κάτω μέλος που είναι ενταγμένο στην διευρυμένη συνεργασία, είναι προφανές ότι θα απαιτείται η φορολόγηση. Το ίδιο και όταν υπάρξει συναλλαγή με ένα ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην ίδια αυτή ζώνη. Θα πρέπει να τεθεί με διαφάνεια το πρόβλημα. Και γι' αυτό είχα εκφράσει τη θλίψη μου, διότι αυτό το αίτημα για ενισχυμένη συνεργασία δεν είχε συνοδευτεί από κάποιο προσχέδιο κειμένο που να δίνει κάποιες ενδείξεις βασικές επ' αυτού. Θα κρίναμε καλύτερα αν είχαν περισσότερα στοιχεία, αλλά προφανώς κάποιοι είχαν συμφέρον να καλλιεργούν ένα κλίμα μυστηρίου. Αυτό δεν είναι κάτι υγιές. Θα μπορούσε να επιφυλάσει άσχημες εκπλήξεις. Παρόλο που έχω ρωτήσεις ε, και προβληματισμό, δεν είμαι αντίθετη. Εγώ θα υποκληθώ στον νόμο της πλειοψηφίας, χωρίς να έχω συγκεκριμένη θέση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα. Και θα πρέπει η πρότασή της να συμπεριλαμβάνει μελέτη αντιχτύπου όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τις διαδραστικές σχέσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών που θα είναι εντός του σχήματος και εκείνων που θα είναι εκτός. Αυτά έχω να πω. Συμφωνώ, όπως είπε και η κυρία εισηγήτρια, με τις ε, δύο συμβιβαστικές ε, προτάσεις που συνέταξε μετά τις προτάσεις μου. Συμφωνώ, αλλά ήθελα να πω ακριβώς τι διακυβεύεται. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις συνέπειες μιας τέτοιας συνεργασίας όσον αφορά τις χώρες που θα είναι εντός και τις χώρες που θα είναι εκτός. Πρέπει ο καθένας να κατανοεί ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι καλή συμβιβαστική τροπολογία. Πιστεύουμε ότι ο FTT θα πετύχει τους στόχους τους αν εισαχθεί σε σφαιρικό επίπεδο ο φόρος αυτός των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα είναι θετικό το παράδειγμα θα είναι αρνητικό, δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε τι έγινε στη Σουηδία. Κατανοώ τους Σουηδούς συναδέλφους. Όταν θέσπισαν τον φόρο αυτό για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στη Σουηδία ήταν επιτυχέστατος νόμος για το Λονδίνο. Μου είπαν ότι οι συναλλαγές που κινήθηκαν προς Δοδίνο δεν, δεν οδήγησαν σε έσοδα για τη Σουηδία. Πρέπει να γίνει σωστή στάθμιση των υπέρ και κατά αυτού του είδους ε, του εγχειρήματο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κλίμπ θα μιλήσει εκ μέρους του κύριου Μοντερούσα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τρεμόσα, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι Καταλανός στην Καταλωνία και έχουν κλέξει μόλις, όπως γνωρίζετε, είναι στην πατρίδα του λοιπόν στην Καταλωνία και τα εκλογικά αποτελέσματα για να τα αξιολογήσει εκεί εξειδικευμένα δεν μπορεί λοιπόν να παραστεί. Δεν μου έδωσε και τίποτα γραπτό ως κείμενο ή έγγραφο. Έτσι πρέπει να αυτοσχεδιάσω λοιπόν παρουσιάζοντας κάποια πράγματα. Να πω το εξή πρώτα. Πρώτα λοιπόν για το θέμα του τέλους ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Πριν από 30 χρόνια, είναι παλιά ιστορία, ξεκινήσαμε με αυτή τη συζήτηση. Και όπως ε, αναφέρεται ότι μπορεί αυτό να είναι χρήσιμο, να χρειαστεί, θα μπορούσε ίσως να ευδοκιμήσει αυτό που προτάθηκε στην, στην αρχή, ε, έδωσε θετικές εντυπώσεις, διότι είπα ότι είναι κάτι το συνετό και λογικό και αν εφαρμοστεί έτσι όπως το στοχεύαμε και με την αρχή της έδρας, δηλαδή ο φόρος να μην μπορεί να διαφύγει όταν κάποιος συναλλάσσεται με αυτόν τον τρόπο και να συμπληρωθεί λοιπόν έτσι με την ε, αρχή του κράτους προέλευσης, πράγμα που θέλει να επιβάλλει το Κοινοβούλιο. Τότε θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Μόνο που καταδείχθηκε εντωμεταξύ ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να εγκρίνουν αυτή την πρόταση πλειοψηφικά και για την αρχή όπως προτάθηκε από την Επιτροπή δεν μπορούν να την υποστηρίξουν αυτή την κατεύθυνση, αυτή την αρχή. Με τον ένα ή άλλο τρόπο θέλουν να μειώσουν σε ένα κανονικό τέλος χρηματιστηρίων που μόνο στα μερίδια και στις ομολογίες και στις μετοχές θα περιορίζεται. Αυτό από πλευρά Σουηδών ε, συναδέφων, π.χ. του Όλε Σμιτ στην ομάδα Άλτε, αυτό το οποίο έγινε στη Σουηδία στο παρελθόν, να συνεχιστεί και να πούμε ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτό το τέλος ε, κλιματοοικονομικών συναλλαγών εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Σουηδία αυτό, τον, ε, αυτό το τέλος όπως το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και αν συναλλάσσονται Σουηδοί στο Λονδίνο να φορολογούνται όχι δεν είχε προβλεφθεί αυτό είχε διαφορετική κατεύθυνση όπως διαμορφώθηκαν όμως τώρα τα πράγματα έχω μεγάλες επιφυλάξεις αυτό το οποίο απέμεινε από τις αρχικές προτάσεις αν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία και να λειτουργήσει καλά πρώτον μόνο κάποιες λίγες χώρες ε, θα συνεργαστούν 11 ή 12 πόσες θα είναι. Αλλά έχουν και διαφορετικές απόψεις αυτές οι χώρες πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το τέλος. Η αρχική προσέγγιση αποδυναμώθηκε ήδη. ποσε τέτοιο τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Από την 1η Αυγούστου στις ε, συμμετοχές στις γαλλικές στο χρηματιστήριο έχουν λέει τέτοιο τέλος. Και ήδη. Λένε οι χωρε πω πρεπει λέει το τελο η αρχικη προσεγγιση αποδυναμωθηκε ηδη λενε οι γαλλοι εχουμε ενα τετοιο τελος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ε δεν είναι βέβαια. Όταν όμως το λένε ότι ισχύει αυτό εκεί και δεν είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν, να τροποποιήσουν δηλαδή αυτό, αυτόν τον φόρο που εισήχθη εκεί και να τον επεκτείνουν, ε, τότε θα έχουμε προβλήματα. Σε σχέση με τα 10 ή 11 κράτη τα οποία είναι πρόθυμα για εμβαθυμένη ε, συνεργασία και συντονισμό, θα έχουμε μεγάλες διαφορές. Δεν θα έχουμε άρρητα εμπόδια. Αντί να ενωστεί η Ευρώπη, θα έχουμε ένα πρόσθετο κατακαιρματισμό ένα πρόσθετο διχασμό και αυτό θα είναι πρόβλημα. Πρώτο σημείο. Δεύτερον, οι χώρε οι οποίε ε, συνεργάζονται, είχαν πει ότι θα συνεργαζόντουσαν, δεν συνεχίζουν αυτή τη συνεργασία διότι σε σχέση με τη χρηματοδότηση για την ε, χρηματοδότηση των ε, αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης λένε ότι αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες ώστε να εισάγονται, να εισπάτονται φόροι. Ε, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι απελπιστική κατάσταση όταν όλοι είναι υπερχρεωμένοι και κάθε τέλος, κάθε εισφορά, κάθε έσοδο είναι ευπρόσδεκτο για αυτούς και γι' αυτό θέλουν να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία χωρίς να ευδοκιμήσει η τελική στοχοθέτηση, δηλαδή ανακούφιση και ελάφρυνση του απλού πολίτη, του φορολογούμενου, ώστε να μπορέσουν να αποσβεστούν ε, οι ζημιές και οι ε, βλάβες που έχουν ε, προκληθεί. Γι' αυτό μπορώ να δώσω δίκιο σε αυτό το οποίο είπε η προλαλή σας, η κυρία Άστριντ Λούλινγκ. Προτού γνωρίσουμε τι συγκεκριμένα με αυτή την τροποποιημένη εισαγωγή αυτού του τέλους, όπως τροποποιήθηκαν τα πράγματα, πώς θα διαμορφωθούν τελικά τα πράγματα και ποιοι θα συμμετάσχουν από πλευράς κατών μελών και ποιοι δεν θα συμμετάσχουν, προτού αποσαφινιστούν όλα αυτά είμαι πολύ επιφυλακτικό όταν πρόκειται για την εισαγωγή αυτού του τέλους. Όταν ακούω ότι ούτως ή άλλως λένε ότι αυτός ο φόρος, αυτό το τέλος δεν θα εισαχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016. Είμαι ακόμα πιο επιφυλακτικός και ολοκληρώνω τελευταία παρατήρηση, δεν γνωρίζω ακόμα και πώς δεν έχει αποσαφινιστεί πώς θα διασφαλίσουμε ότι το τέλος αυτό θα εισπράτεται ως φόρος με ομαλό και τακτικό τρόπο και πώς θα εμβάζεται. Πώς, διότι πολλές χώρες οι οποίες δεν θα συμμετάσχουν αλλά πρέπει να εισπράττουν φόρους ε, τέτοιου είδους έσοδα με την αρχή του κράτους προέλευσης. Πιθανότατα λοιπόν αυτές οι φορολογικές ε, διοικητικές υποθέσεις ε, θα πρέπει πρώτα να έχουν αποσαφινιστεί πρωτού προχωρήσουμε. Δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Έχω λοιπόν σοβαρές επιφυλάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Η κυρία είναι εκ μέρους των Πρασίνων έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ τον εισηγητή που τα κράτησε πιο απλά τα πράγματα, σε ένα απλούστερο πλαίσιο, σημαντικό σε αυτή τη φάση. Και μας υπενθυμίζει ότι διαδικαστικά είναι θέμα που αφορά τη συνένεση. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα ουσίας, είναι σαφές αυτό, είναι μια πολιτικής μορφής πρόταση. Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα ουσίας. Αλλά πάλι θέλω να απευθύνω έκκληση εδώ στην Άλντε και στο ΕΛΚΑ που τοποθετήθηκαν και ανέφεραν σε επιφυλάξεις τους να επανεξετάσουν και να δουν είναι ο ρόλος ε, του Ευρωκοινοβουλίου να αναχαιτήσουν, να σταματήσουν 11 κράτη-μέλη και τουλάχιστον ε, νομίζω ότι θα έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις και αυτές οι χώρες που είναι εκτός και δεν θέλουν να συμμετάσχουν υποθέτω ότι τα Υπουργεία Οικονομικών τους έχουν την ικανότητα να υπολογίσουν τι θα μπορούσαν να εισπράξουν και τι όχι. Αν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κάπως το Κοινοβούλιο θα εκφράσει ενστάσεις, ή θα είχε αντιρρήσεις, νομίζω αυτό θα ήταν πραγματικά παράλογο και εξοργιστικό. Να το αποσαφηνίσω αυτό. Δεν το μπορώ να το φανταστώ. Το κάναμε αυτό σε Ευρωβουλή. Για φανταστείτε μια κατάσταση να εκφράζει ανησυχίε στο Ευρωκοινοβούλιο και να λέει δεν είναι έτοιμο να δώσει τη συνένεση, ενώ το σύνολο των κρατών στο Συμβούλιο είναι να, έτοιμα να προχωρήσουν και π.χ. για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει κάποιες ε, ενστάσεις, θέλω να απευθύνω έκκληση να τα επανεξετάσετε αυτά να τα λάβετε όλα υπόψη. Δεν είναι δική μας δουλειά στην Ευρωβουλή να επιβραδύνουμε τις διεργασίες. Από την άλλη πλευρά θα έπρεπε να επιτρέψουμε σε αυτές τις χώρες να προχωρήσουν αν αυτό επιθυμούν. Και τώρα επί της ουσίας για να σχολιάσω κάποια πράγματα αν επιτρέπετε. Ένα από αυτά είναι ότι για την ενιαία εσωτερική αγορά και η κυρία Λίλινγκ μαζί με τον κύριο Κλίντς αμφότεροι ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις για τις χώρες εκτός και θα μπορούσε να έχει επιπτώσει σε αυτή η πρωτοβουλία για την εσωτερική αγορά. Μία παρατήρηση. Κατακαιρματισμό υπάρχει ήδη σήμερα λοιπόν. Δεν θα δημιουργήσει αυτή η πρόταση περαιτέρω κατακαιρματισμό. Έχουμε σήμερα ήδη 8 χώρε με ένα είδο τέλο τέτοιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εμεί θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο τέλο χρηματοοικονομικών συναλλαγών όπου περισσότερε από 11 χώρε θα συμμετάσχουν και θα περιοριστεί ο κατακαιρματισμό. Διότι ο κατακαιρματισμό υφίσταται ήδη σήμερα αυτό, ε, αυτού του θέματο σήμερα και είναι σημαντικό επιχείρημα να λάβουμε υπόψη αυτό. Δεύτερον, για τις χώρες εκτός είναι αρνητικό, είναι δική τους υπόθεση θα έλεγα να αξιολογήσουν τα πράγματα οι χώρες αυτές και να δουν τι θα κάνουν. Όταν τα συζητούσαμε προηγούμενα πάντα είχαμε τη λογική ότι θα ήταν κακό από εκείνες τις 27 χώρες που το υιοθέτησαν και θα ήταν καλό λέει για όλες τις άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ανα, ανατράπηκε αυτό το επιχείρημα, ισχύει λέει διαφορετικά, δεν μπορώ να κατανοήσω πλέον τη λογική των πραγμάτων. Είναι δυσνόητο για τη Σουηδία η Σουηδία είναι το εσωτερικό υπόδειγμα, παράδειγμα, τι να μην κάνουμε, τι να αποφύγουμε. Φυσικά μπορεί να σχεδιάσει κανείς ένα αρνητικό τέτοιο τέλος συναλλαγών. Κάθε είδος τέτοιου τέλους δεν μπορεί να είναι, όλα, δεν μπορεί να είναι πάντα ιδανικό. Αυτό το οποίο σχεδιάστηκε λυπούμε, υπάρχουν και Σουηδοί συνάδελφοι, ήταν πολύ πενιχρό και δεν, είχε, δεν ήταν καλά σχεδιασμένο. Και εδώ για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σχέση με τη Σουηδία, ας μάθουμε, συνεργάζουμε τα συμπεράσματα από αυτά, αλλά ας δούμε και το τι πρέπει να γίνει για χώρες που υπάρχουν και έχουν ένα τέλος τέτοιας χρηματοοικονομικής ίσπραξης ε, ε, επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών, είναι το θέμα του πώς τα σχεδιάζει κανείς για να είναι αποτελεσματικό αυτό. Είμαι ικανοποιημένη, χαίρομαι για το ότι τα πράγματα εξετάζονται όπως ε, πρότεινε το Ευρωκοινοβούλιο για να συνεισφέρουμε στην αρχή έκδοσης. Η αρχή έκδοσης να προσθέσει τεθεί αυτή όσον αφορά την λειτουργία αυτού του τέλους ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Να το δούμε αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει έτσι για να προχωρήσουμε. Και τέλος, θα έλεγα, ίσως είναι η χρονική στιγμή που θα έπρεπε ιδεολογικά να μην διεξάγουμε ιδεολειπτικά τη συζήτηση, να σκεφτούμε το ρόλο μας ως Ευρωκοινοβούλιο σε μια διευρυμένη διαδικασία. Θα έχουμε ευκαιρίες να επανέλθουμε στο μέλλον επί της ουσίας συζητώντας αυτή την πρόταση όταν θα έχει προχωρήσει, όταν θα έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε την συνένεσή μας για αυτή τη διαδικασία για να προχωρήσει. Και μπορεί νομίζω αυτό να μας προχωρήσει στα θέματα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τουρούνεν. Ο κύριος Στράγεχ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει ο κύριος Στρέιτσεκ. Ουσιαστικά όταν παρεμβαίνω χρησιμοποιώ την αγγλική γλώσσα σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά μια και κάνουμε λόγο για αυτό το συγκεκριμένο εξειδικευμένο θέμα, φοβούμε ότι θα έπρεπε να ε, μιλήσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό ε, με τρόπο ώστε να μην θεωρεί κανείς ότι το Λονδίνο εκπροσωπείται και ότι κάποιος μπορεί να ε, έχει μια τέτοια θέση. Γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω στη δική μου μητρική γλώσσα. Και έτσι για να αποδείξω ότι το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχει και άλλους οπαδούς. Ε, έχει ευρωβουλευτές από άλλες χώρες που θεωρούν ότι αυτή η αρχή είναι κάπως αντιφατική αυτή η προσέγγιση για να το εκφράσω κατεφημισμών. Δεν έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες ή προτάσεις και έτσι δεν πρόκειται να τοποθετηθώ επ' αυτών μακρηγορώντας. Θα ήθελα όμως κάποια λίγα σχόλια, κάποιες λίγες παρατηρήσεις να κάνω προς την κυρία Τουρούνεν. Η κυρία Τουρούνεν τι συνέστησε. Συνέστησε να μην είναι ιδεολειπτική και ιδεολογική συζήτηση, αν κατάλαβα καλά. Εντάξει, ναι, προφανώς. Λοιπόν, σωστό αυτό. Όμως όταν κάνουμε λόγο για φόρους, για την εισαγωγή και υλοποίηση νέων μορφών φόρων, δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια προσέγγιση. Υπάρχουν άτομα που, πρέπει να που λένε ότι πρέπει να αποφασιστεί και να εισαχθεί αυτό. Άλλοι λένε να μην εισαχθούν νέοι φόροι και τέλη. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος ούτε τραπεζικών ιδρυμάτων ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Αν είναι τόσο εύκολο μόνο να κατηγορούνται οι τράπεζες ως η μόνη πηγή, το μόνο αίτιο όλων αυτών των προβλημάτων, τότε θα ήταν απλή η κατάσταση των πραγμάτων στην οικονομική ζωή και θα μπορούσαμε με απλούστερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αλλά δεν πιστεύω ότι έτσι απλά μπορούμε συλλήδιν να κατηγορούμε ισοπεδωτικά τις τράπεζες ως μόνες υπέτειες. Και τώρα σε σχέση με μια ήπια μορφή τέτοιου φόρου ή μέσα στο συνολικό φορολογικό πλαίσιο η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη από να είχαμε το θέμα αυτό για να αναλυφθούν τέτοιου είδους ε, μέτρα για την διαχείριση. Δεν πιστεύουμε ότι νέα, ε, νέοι πόροι, νέα χρήματα μπορούν να εξευρεθούν που κανείς δεν είχε φανταστεί κατά το παρελθόν. Αυτά τα χρήματα θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των καταναλωτών μας. Να πιστεύει κανείς ότι το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα είναι μια πηγή άντλησης κονδυλίων από νέες πηγές δεν έσταθεί. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους νέο χρήμα το οποίο να πέφτει στα χέρια σας με ένα μαγικό ραβδί. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να στεφθεί με επιτυχία ως εγχείρημα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και θεωρούμε ότι αν εισαχθεί κάτι τέτοιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να είναι επιζήμιο, να έχει επιζήμιες επιπτώσεις όσον αφορά την οικονομία. Αν κατάλαβα καλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ίδια διαρωτάται και θέτει αυτό το ερώτημα και έκρουσε κόδωνα κινδύνου κατά δυνατόν ενδυνάμει τέτοιων αρνητικών επιζήμιων επιπτώσεων λόγω εισαγωγής ενός τέτοιου φόρου χρηματικών συναλλαγών. Ε, συμπεράσματι, η, κατάσταση, η τοποθέτησή μας πλησιάζει εκείνη κάποιων τροπολογιών που κατατέθηκαν από κάποιους ευρωβουλευτές, π.χ. του κυρίου Χεκμάρκα, π.χ. του κυρίου Σμιτ. Και πιστεύω ότι ο συνάδελφος Κλίντς επίσης ε, έχει συνυπογράψει και εκείνος ε, τέτοιες προτάσεις. Έχουμε προσεγγίσει λοιπόν αυτές τις ε, προτάσεις, αυτές τις τροπολογίες, προσεγγίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις αυτών των συναδέφων. Τώρα, Συμπερασματικά, αν καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση, αυτό δεν θα σημαίνει ότι είμαστε αρνητικοί εναντίον όλων των προτάσεων. Κάποιες από αυτές θεωρούμε θετικές. Ευχαριστώ. E Τώρα, ο κ. Κλούτε θα μιλήσει εκ μέρους της Μαρίζα Ματίας. Μάλιστα. Θα πρέπει να ζητήσω συνα... Ε, συγγνώμη από τη συνάδελφα. Δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα το πρωί και με παρακάλεσε στη θέση τη να πω κάποια πράγματα. Μου σημείωσε κάποια πράγματα τα οποία θα σα τα διαβάσω από πλευρά κειμένου θα ήθελα όμως κάποιες δικές μου προσωπικές παρατηρήσεις να κάνω πρώτα. Και επισημάνθηκαν οι επιφυλάξεις που υπάρχουν όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της εισαγωγής ενός τέτοιου τέλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η κυρία Άστριντ Λούλινγκ ε, επεσήμανε τα προβλήματα όπως υπάρχουν. Θα ήθελα και πολιτικά και ιδεολογικά, ιδεολογικά να πω τα εξή. Αυτές τις επιφυλάξεις θα επιθυμούσα να τις ακούγαμε πριν από τις μισθολογικές περικοπές ε, που επιβλήθηκαν στις χώρες που αντιμετωπίζουν την κρίση σήμερα, την ε, Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, δεν διαρωτήθηκαν διαμακρών ε, τι, ποιες επιπτώσεις αρνητικές θα υπήρχαν, απλώς επιβλήθηκαν αυτές οι περικοπές. Εδώ όμως για, το, για την εισαγωγή του τέλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών συζητούμε και μάλιστα συζητούμε διαμακρών ε, επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται που λόγω των περικοπών ε, έχουν πληγεί πολύ σημαντικά θα ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους ε, επιχειρήματα. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κλίνς ε, και για το Συμβούλιο. Καταρχήν το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο είναι γνωστό για τέτοια πράγματα. Όταν πρόκειται για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενιαία εσωτερική αγορά, το φρένο, η αναχέτηση προέρχεται από το Συμβούλιο. Είναι προφανές τουλάχιστον εγώ θα ήθελα να το καταστήσω σαφές αυτό προσωπικά ο ίδιος. Και για μένα αυτό αποτελεί λόγο για να πούμε ότι θα έπρεπε να δώσουμε συνέχεια σε αυτήν την πρωτοβουλία. Γιατί διαφορετικά θα καταλήγαμε και μπορεί κανείς αυτό να το ερμηνεύσει ως ε, παρελκυστική τακτική ε, για επιβράνηση, για καθυστέρηση από το Συμβούλιο και όλα αυτά να χαθούν μετά στο τέλος, να μην οδηγήσουν πουθενά. Γι' αυτό πρέπει πιστεύω να κάνουμε κάτι για τους πολίτες, τους απλούς καθημερινούς ε, πολίτες, τους κοινούς θνητούς και να μην αφήσουμε να παρέλθει και να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να δραχθούμε τη ευκαιρία να κάνουμε κάτι υπέρ των ε, φορολογουμένων. Θα σα διαβάσω το κείμενο τη Μαρίζα στα αγγλικά. Μου ε, κατέγραψε εδώ κάποια πράγματα σε κάποιε αράδε. Λοιπόν, αγγλικά. Η εισαγωγή του φόρου του τέλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των οικονομικών αγορών και για την δικαιότερη κατανομή για την εισφορά της χρηματοδότησης των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι ε, που θα έχει θετικές επιπτώσεις και θα μειωθεί η μεταβλητότητα, ο ευμετάβλητος χαρακτήρας ε, των χρηματοοικονομικών συναλλαγών όπως υφίστανται σήμερα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, υπάρχει πολύ ήπιος, ήπια δομή όσον αφορά την πρόταση και θα πρέπει να στοχεύουμε στην ίδια την, τον ίδιο τον πυρήνα. Είναι ένα όμως σημαντικό βήμα, πρώτο βήμα, ώστε να μπορέσουν οι αγορές να εξυπηρετήσουν την οικονομία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτός ο ευκταίος στόχος σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα έπρεπε να συνοδεύεται με την ε, επιστράτευση των ε, εσόδων για να υποστηριχθεί η αηφορία και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα έσοδα από τον, το τέλος ε, της ε, συναλλαγής αν αυτά από τον προϋπολογισμό τότε δεν θα δώσουν τη δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι ατυχές λοιπόν ότι αυτό το κείμενο αυτό δεν εισάγεται στο κείμενο σε σχέση με την ΕΕ. Προφανώς κάποιες ε, κυβερνήσεις ε, αντιδρούν ταχύτατα όταν έρχεται η ε, στιγμή να ε, επιβληθούν κάποιες κυρώσεις, κάποιες περικοπές σε σχέση με τους μισθούς των Ευρωπαίων πολιτών και δεν είναι πρόθυμες με τον ίδιο ταχύ ρυθμό να ε, επομιστούν τις ευθύνες τους σε σχέση με μια άλλη κατεύθυνση. Και για την εισαγωγή ενός τέτοιου τέλους ε, το ότι όπως λένε κάποιοι θα αναγκαστούν ε, εταιρείε να μετεγκατασταθούν από την Ευρώπη είναι αξιοπρόσεκτο ότι τέτοιου είδου επιχειρήματα αναφέρονται από χώρες ε, του, της Ενωμένης Ευρώπης όπως ε, το, από το Ενωμένο Βασίλειο για παράδειγμα που έχει μια ξεχωριστή τοποθέτηση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Η εφαρμογή αυτή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να δώσει μέσα σε ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο θετικές ε, επιπτώσεις. Το πλήρες ε, δυναμικό όμως ε, μπορεί να αναπτυχθεί και να επιτευχθεί όταν πανευρωπαϊκά θα μπορέσει να εισαχθεί σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Θα πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εξυπηρετείται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά τα έσοδα. Έτσι να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίζουμε σήμερα, μιλώντα ε, και για αλληλεγγύη στην Ευρώπη, σημαντικό είναι μετά από τα λόγια να περάσουμε στι πράξεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό είναι το κείμενο της Μαρίζα Ματία στα αγγλικά, όπω μου το σημείωσε. Και τελευταία τώρα θα ήθελα να υποβάλω σε σχέση με την τροπολογία H, την τελευταία πρόταση όπου λέγεται διευρυμένη συνεργασία, επίσης μπορεί να δώσει θετικά ένα θετικό παράδειγμα για την εισαγωγή του τέλους χρηματοοικονομικής συναλλαγής σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι το κείμενο και σε σχέση με την διαγραφή δεν μπορώ να κατανοήσω πρέπει να πω γιατί γίνεται αυτό, γιατί ζητείτε να μην, αν θα μπορούσε να ζητηθεί να μην διαγραφεί από πλευρά εισηγητού αυτό, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε υστερότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Κάποιο θέλει να παρέμβει από τους ευρωβουλευτές τα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Κύριε Βάγκμαν έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις συζητήσεις και αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Κοινοβούλιο και έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο γύρω από το θέμα αυτό. Ήταν πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Τρία σημεία για την κριτική και τον σκεπτικισμό που ακούστηκε εδώ πρώτον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πρόταση αυτή επί της ουσίας θα διαιρέσει την Ευρώπη. Όχι, θα ενισχύσει την διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ενίας αγοράς και θα γίνουν καλύτερα σεβαστές οι ισχύουσες ρυθμίσεις, γιατί θα υπάρχει καλύτερο νομικό πλαίσιο. Δεύτερον, δεν σύμφωνα με αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ σχετικά με την υπερεδαφικότητα. <clears throat> τα πιστοτικά ιδρύματα, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μη συμμετεχούσων χωρών είναι μια αρχή η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Τα ιδρύματα αυτά θα πρέπει να πληρώνουν το φόρο εκεί όπου δραστηριοποιούνται εφόσον η νομική ρύθμιση το επιβάλλει. Το θέμα δεν είναι μόνο από πού προέρχονται ας πούμε κάποια προϊόντα, αλλά το θέμα είναι με ποιον γίνεται η ε, συναλλαγή των προϊόντων αυτών. Τώρα, ο έλεγχος και η επιβολή στο εσωτερικό των κρατών μελών, κάτι τέτοιο είναι εφικτό θα έλεγα, για να μην πω εύκολο. Ίσως να είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα στις μη συμμετέχουσες χώρες. Σας συμμεριζόμουν την ανησυχία σας. Αν λειτουργούσαμε με ένα παλαιότερο σύστημα στα πλαίσια του οποίου δεν υπήρχε διαφάνεια και οι θύρες ήσαν κλειστές. Τώρα όμως η αγορά είναι αρκετά διαφανής. Έχουμε επιπλέον νομικά μέσα στον τομέα των κανονισμών των χρηματαγορών που θα καταστήσουν εύκολο το να ορίζουμε το ποιοι θα πρέπει να πληρώνουν και πόσο και έτσι οι αρχές ε, ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν τις πληρωμές από αυτούς που δεν έχουν πληρώσει. Τέλος για την μελέτη των επιπτώσεων, όπως είπαμε εμείς έχουμε κάνει μια τέτοια μελέτη στα πλαίσια της αρχικής πρότασης, έχουμε στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύσει συμπληρωματικά στοιχεία και εσωτερικά τώρα προσπαθούμε να δούμε τι αναλύσεις μπορούμε να κάνουμε και τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε Έχουμε επίσης επαφή και με την νομική υπηρεσία και με άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει μια ομάδα ε, επεξεργασίας και ελέγχου της μελέτης των επιπτώσεων η οποία ήδη από αύριο δραστηριοποιείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την πρότασή της επί της ουσίας θα καταθέσει και ένα κείμενο το οποίο θα αναλύει τις ε, ε, επιλογές πρακτικές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε ε, και θα υπάρξει και το λεγόμενο CIA, δηλαδή συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων. Να σας διαβεβαιώσω ότι σύμφωνα πάντως με τα πρώτα ευρήματα δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις είτε στις συμμετέχουσες χώρες είτε στις μη συμμετέχουσες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Μπάγκμαν. Η κυρία Ποδηματά για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ελληνικά ε, στη δευτερολογία μου, αν ε, ε, είναι εντάξει αυτό με όλους. Θέλω πρώτα να επισημάνω το, το εξής για την συζήτηση που έγινε. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό σε αυτήν την φάση που διανύουμε και είναι ένα από τα πράγματα που υπογραμμίζω κατεξοχήν και στο εσωτερικό της χώρας μου και στο ευρωπαϊκό επίπεδο ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, στο μέσο αυτής της κρίσης που είναι κρίση αξιοπιστίας να κάνουμε όλη μια προσπάθεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι ε, έχει δώσει το παράδειγμα σε πολλές περιπτώσεις προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς στο λόγο μας και επίσης ε, να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στο λόγο μας και στις πράξεις μας. Ε, το λέω αυτό πρώτα απ' όλα για να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει με μεγάλη πλειοψηφία μια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, στην Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά επί της ουσίας όταν υποβληθεί η αναθεωρημένη και προσαρμοσμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αλλά ταυτοχρόνως να συγκρατούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ε, το πλαίσιο της τοποθέτησης που πριν από έξι μόλις μήνες ε, είχε υπάρξει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό δεν σημαίνει με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτηση μιας θέσης ότι αυτοί που έχουν επιφυλάξεις ή που είναι πολέμοι δεν έχουν το, το απόλυτο δικαίωμα να διατηρούν τις δικές τους απόψεις. Ε, υπάρχει όμως νομίζω και εκεί μια υποχρέωση να είμαστε ε, συνεπείς με την επιχειρηματολογία που αναπτύσσουμε. Και θέλω να θυμίσω ότι η πολέμοι του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εκείνοι που είχαν ισχυρές επιφυλάξεις στις συζητήσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, χρησιμοποιούσαν κυρίως και κατεξοχήν ένα επιχείρημα που ήταν ο κίνδυνος της φυγής ε, συναλλαγών και ε, χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων εκτός της ε, ευρωπαϊκής επικράτειας, διότι εκείνη την περίοδο μιλάγαμε για φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το βασικό επιχείρημα λοιπόν ήταν ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου φόρου θα οδηγούσε σε φυγή συναλλαγών ή και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας προς προορισμούς με πολύ ευνοϊκότερο ε, φορολογικό καθεστώς από αυτό που θα εισήγετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τώρα λοιπόν που εξετάζουμε την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, που έχουμε 11 κράτη-μέλη που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση και την επιθυμία να προχωρήσουν στην εφαρμογή αυτού του φόρου, ε, εγκαταλείπεται αυτό το επιχείρημα και έχουμε πάλι ένα επιχείρημα που εκφράζεται κυρίως από αυτούς που δεν εντάσσονται στους 11 δεν θα εφαρμόσουν δηλαδή ε, το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όχι πλέον με επίκεντρο ε, τον κίνδυνο φυγής συναλλαγών ε, ή και ιδρυμάτων εκτός της επικράτειας όπου θα ισχύσει ο φόρος, αλλά τον κίνδυνο να υπάρξουν επιπτώσεις σοβαρές, το της που λέμε, σε αυτούς οι οποίοι δεν θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου. Άρα λοιπόν η ε, εκείνα τα κράτη-μέλη που θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου σε πρώτη φάση δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Υποθέτω ότι ουδής το πιστεύει αυτό, ότι οι κυβερνήσεις και οι Υπουργοί Οικονομικών των 11 δεν ε, αξιολογούν σωστά ε, τις επιπτώσεις που θα έχει ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρωτίστως στη δική τους επικράτεια είτε όπως σημείωσα και στην αρχή θεωρούμε ότι θα είναι τόσο επιτυχής ε, η εφαρμογή του φόρου αυτού, σε αντίθεση με ό,τι λέγαμε πριν από λίγους μήνες, ώστε θα προκύψει κόστος και μάλιστα ε, σημαντικό, αξιοσημείωτο, δυσβάστακτο, θα προκύψει κόστος σε αυτούς που δεν θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του φόρου. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι μια ε, υπερβολή και είναι σε, αναντιστοιχεία με την επιχειρηματολογία που είχε αναπτυχθεί από τους ενάντιους το προηγούμενο διάστημα και το επισημαίνω αυτό ε, ε απλώς για να υπογραμμίσω ότι ε, μπορούμε να έχουμε ε, απόψεις ισχυρές υπέρ ή κατά του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό είναι ασφαλώς θεμητό αλλά θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς την επιχειρηματολογία που ε, αναπτύσσουμε. Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα πιστούν ε, από, την, από τα ωφέλη που μπορεί να προκύψουν ε, από την εφαρμογή αυτού του φόρου έτσι και αλλιώς. Ε, το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ε, δεν έχουμε ανάγκη από άλλο έναν φόρο. Είμαστε σε μια, αναφέρομαι κυρίως σε μια επισήμανση που έγινε από την πλευρά του, ε, συναδέλφου του Wolf Klintz στη συνέχεια από τον συνάδελφο τον Στρέτσεκ είμαστε σε μια διαδικασία υπερφορολόγησης υπάρχουν υπερφορολογημένοι υπερχρεωμένοι και δεν μας χρειάζεται ένας ακόμα φόρος ο οποίος θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ε, θα επιφέρει νέα επιβάρυνση. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι είμαστε υπερχρεωμένοι, υπάρχει υπερφορολόγηση, αλλά πού υπάρχει υπερφορολόγηση. Η υπερφορολόγηση υπάρχει στον, στους ανθρώπους της εργασίας και η υπερφορολόγηση υπάρχει στην παραγωγική ε, οικονομία. Λοιπόν, είναι ζήτημα ε, ενός δικαιότερου επιμερισμού των βαρών, αν θέλετε. Το έχουμε επισημάνει αυτό πολλές φορές στη διάρκεια αυτής της τριετίας. Δεν είναι ζήτημα, κύριε Στρέτσετ, εκδίκησης των τραπεζών και ουδής δεν θεωρεί ότι οι τράπεζες είναι οι μοναδικέ πέτειες. Άλλωστε, θέλω να θυμίσω ότι το βάρος της κρίσης κατά βάση εθνική εθνικοί το σηκώνουν σήμερα, ε, δεν το σηκώνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη σωτηρία του επιστρατεύτηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ ε, τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, είναι απλώς ένα ζήτημα δικαιότερου επιμερισμού του κόστους της κρίσης και δικαιότερου επιμερισμού των βαρών της φορολόγησης. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει αυτό το καθεστώς της υπερφορολόγησης που επιβαρύνει όμως στον κόσμο της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, ε, ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα συμβάλλει σε αυτόν τον δικαιότερο επιμερισμό του κόστους και του βάρους της, ε, της φορολόγησης. Τέλος, ε, τελειώνω. Τέλος, είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη φόρου φορολόγησης χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διάφορα κράτη-μέλη σήμερα και μεταξύ των 11. Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Γαλλίας, μα ακριβώς και η αρχική πρόταση ε, που στόχευε στην εισαγωγή του φόρου σε επίπεδο 27 και η σημερινή πρόταση στη βάση του κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε απόφαση μεταξύ των 27 με ομοφωνία στοχεύει ε, στην αντιμετώπιση αυτού του, του κατακαιρματισμού που υπάρχει σήμερα στη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη και στην μεγαλύτερη εναρμόνιση, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι προ όφελο τη εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρούμε ότι υπηρετούμε την ε, εσωτερική αγορά ε, με μεγαλύτερη συνέπεια και επιτυχία ε, ανεχόμενη ή ενθαρρύνοντας αν θέλετε την παράταση αυτού του απόλυτου κατακαιρματισμού. Ε, η εισαγωγή αυτού του φόρου πρώτα απ' όλα μεταξύ των 11 θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα εναρμόνισης που οπωσδήποτε θα αποβεί ε, προς το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών. Τέλος, επειδή ρώτησε κάτι συγκεκριμένο, ο Γιούργεν ε, σε ό,τι αφορά την μία από τις δύο συμβιβαστικές τροπολογίες και την αφαίρεση του όρου θετικό παράδειγμα. Γιούργεν, η γνώμη μου είναι ότι όταν λέμε θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα εννοείται ότι είναι θετικό. Αφαίρεσα τη λέξη θετικό ε, για να καλύψω την ε, ε, τροπολογία που είχε υποβάλει η Astrid λούλινγκ αφήνοντας το περιθώριο να ερμηνεύσει ο καθένας, παρά ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι όταν λέμε χρησιμεύει ως παράδειγμα είναι θετικό παράδειγμα και όχι αρνητικό, αλλά σε μια προσπάθεια ε, να σηματοδοτήσουμε την ευρύτερη δυνατή ε, ε, συνένεση με δεδομένο ότι μιλάμε για μια έκθεση που στοχεύει στο να δώσει την, άδεια, την έγκριση, τη συνένεση του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας. Very much indeed, Mrs. Podimata. I remind you, uh, Mrs. Luling, we are out of... Ευχαριστώ κυρία Παδηματά. Ένα λεπτό κυρία Λούλινγκ μόλις. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να πω ότι εκπλήσωμαι από την, ε, το αγαθό της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στις υπόλοιπες χώρες. Μία ερώτηση. Στην πρώτη ε, ε, έκθεση την, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ποδηματά και που είχε γίνει δεκτή με πλειοψηφία στην Ολομέλεια, είχαμε κάνει την πρόταση να εξαιρέσουμε τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Είχα ζητήσει επίσης να μην εφαρμοστεί ε, σε τέτοιου είδους οργανώσεις ο φόρος αυτός ο χρηματοοικονομικός ούτε στα usage γιατί είναι κάτι τέτοιο που θα δημιουργήσει πλημμυρίδα αρνητικών επιπτώσεων. Τώρα βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει εκ νέου να συμπεριλάβει ε, στο πεδίο εφαρμογής ε, του ε, φόρου αυτού και τα usage. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν πράγματι εμένει σε αυτό ή όχι. Ο κύριος Μπάγκμαν, κυρία Λούλινγκ δεν είναι εδώ, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχει φύγει πλέον. Γίνεται συζήτηση εκτός μικροφώνου με την κυρία Πόδηματά και την κυρία Λούλινγκ. Λοιπόν, γνωρίζετε Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Ελπίζω κατά τη διάρκεια της ε, ε, ολομελίας του μηνός Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Και τώρα θα περάσουμε στο θέμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Ο κ. Ντεμπάκερ έχει τον λόγο από πλευράς των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που επέδειξαν. Να ευχαριστήσω και τους Σκιώδης για τις τεράστιες προσπάθειες τις οποίες έχουν ήδη κάνει στον συγκεκριμένο τομέα. Άνω των 140 τροπολογιών έχουν κατατεθεί που καλύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος προχώρησα στην επεξεργασία των λεγόμενων συμβιβαστικών προτάσεων Σχετικά με τις ε, τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το κείμενο ε, αναγνώσιμο και ταυτόχρονα κατανοητό. Γι' αυτό δεν ε, δεχθήκαμε τις τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, να μην συμπεριλάβουμε θέματα τα οποία ανήκουν σε αρμοδιότητες άλλων επιτοπών και όπως σας είπα θα θέλαμε η πρόταση αυτή να παραμείνει συνοπτική και διαφανής. Στόχος μας είναι να δώσουμε κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με συγκεκριμένες προτάσεις. Ταυτόχρονα θα θέλαμε να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβασή του στη χρηματοδότηση, αλλά όχι να καταστήσουμε την πρότασή μας σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο με χιλιάδες διαφορετικά θέματα. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε ένα τελικό κείμενο γραφειοκρατικό που δεν είναι στι προθέσεις μας. Συνοπτικά τώρα, τα βασικά χαρακτηριστικά του εγγράφου το οποίο σας ε, καταθέτω. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει μια λύση ενός μεγέθους για όλους Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές, εθνικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Φυσικά, σκελετός της οικονομίας μας είναι οι μικρομεσαίες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δημιουργήσουμε ένα επιπλέον επίπεδο γραφειοκρατικών εμποδίων μέσω των νέων κανόνων και ρυθμίσεων. Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το ε, επιχειρηματικό κλίμα μέσω των βασικών αρχών τις οποίες προτείνουμε. Γνωρίζουμε τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είδαμε ότι οι τράπεζες πέρασαν από μεγάλες καταιγίδε, από ισχυρές καταιγίδε και επηρέασαν αρνητικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν δυνατότητες εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα φορολογικά, θα πρέπει να υπάρξουν επίσης δυνατότητες για την βελτίωση του επενδυτικού χαρακτήρα των ε, of entrepreneurship. Ε, entrepreneurs sometimes lack basic knowledge of finance, accounting, business των ε, καταθέσεων σε ταμιευτήρια και γενικότερα των λογαριασμών από ταμιεύσεις. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι η βελτίωση της διαφάνειας για τους επιχειρηματίες να γνωρίζουν σαν παράδειγμα γιατί έχει απορριφθεί μια αίτησή τους για χρηματοδότηση ή γιατί είναι ή δεν είναι εφικτή η πρόορη επιστροφή των ποσών που έχουν δοθεί. Ε, νομίζω αυτό θα βοηθήσει το κλίμα νομίζω ότι στα πλαίσια της συνάντησης που θα οργανώσουμε το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο να καταλήξουμε σε μια τελική διατύπωση και θα συνεργαστώ και με τους υπόλοιπους σκιώδεις έτσι ώστε η συμφωνία να είναι τελικά θετική. Ευχαριστώ Φίλιπ. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για τη συνεργασία που τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε και που οδήγησε στο, στις συμβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν να μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω δεν έχουμε μεγάλες πλέον διαφορές σε σχέση με αυτή την έκθεση μεταξύ μας. Πολύ σύντομα, εκείνα τα σημεία θέλω να αναφέρω που για μας έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα και που όμως σε μεγάλο βαθμό λαμβάνονται υπόψη στις συμβαστικέ τροπολογίε από την άλλη πλευρά. Αφενό αυτό αναφέρεται από τον συνάδελφο κιόλα το θέμα τη αναλογία ή αναλογικότητα του συσχετισμού μεταξύ τραπεζών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ σίγουρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Όμω εφιστούμε την προσοχή και επισημαίνουμε ότι εξακολουθούν να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι τράπεζες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κατά τούτο λοιπόν απορρίπτουμε προτάσεις. Απορρίπτουμε προτάσεις που στοχεύουν εδώ να εισαχθούν μηχανισμοί που θα επιβάλλουν στις τράπεζες να εγκρίνουν δάνεια και να παρέχουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει η ίδια η απόφαση της τράπεζας να είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα αν θα δίνει ή όχι τέτοια δάνεια. Και έτσι πρέπει να βελτιωθούν λοιπόν τα πράγματα. Μετά επισημαίνουμε και κάτι άλλο, ότι αυτή η κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη, είναι αυτονόητο ότι έχει δραστικές, πολύ μ, ριζοσπαστικές επιπτώσεις σε σχέση με την έγκριση και χωρίση δανείων και πιστώσεων. Στην Ευρωβουλή πολλές φορές γίνεται λόγος για το spread, την διαφορά των επιτοκίων όσον αφορά την κρατική υπερχρέωση, αλλά και σε σχέση με την έγκριση δανείων για την ε, Ευρώπη. Σήμερα Υπάρχει σημαντικό σπρέτ, σημαντική διαφορά μεταξύ επιτοκίων στα διαφορετικά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οδηγεί στο ότι να στρεβλώνεται η ενιαία εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερα όσον αφορά και τις διασυνοριακές μεθοριακές περιοχές που πλήττονται μια και έχουμε διαφορετικές χώρες και που σε πολύ μικρό ε, γεωγραφικό χώρο υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια που ισχύουν και επιβάλλονται. Ένα άλλο θέμα στο οποίο σε σχέση με την Ευρωβουλή θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η επίπτωση των ρυθμίσεων στο τραπεζικό τομέα όσον αφορά την έγκριση δανείων και πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πιο δραστικές επιπτώσεις απορρέουν από την εφαρμογή του ΣΕΕΝΤΕΡΦΙΡ 4 των πλαισίων δηλαδή που συζητούμε είναι σαφές ότι σε σχέση με τις συμφωνίες της ε, Βασιλείας όσον αφορά την αύξηση του ιδίου ε, κεφαλαίου από κάπου πρέπει να αντληθούν αυτά τα ίδια κεφάλαια ώστε τα χρήματα ε, τα οποία θα διατίθενται για τα δάνεια ε, όταν υπάρχει συρρήκνωση να μπορούν να καλύπτονται. Πρέπει υπό αυτή την πτυχή να καλύψουμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι οι πλατφόρμες εγγυήσεων. Υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχουν παιδεία, στο το πω έτσι, εγγυήσεων, εγγυήσει και εχέγγυα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως πλατφόρμες που λειτουργούν θετικά και μπορεί να αποδειχθεί ότι τέτοιες ε, πλατφόρμες μπορούν να ε, συνεισφέρουν ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα σε σχέση με τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τέτοιες πλατφόρμες εγγύσεων. Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να προβληματιστούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες, τέτοια πεδία εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα δάνειά τους. Σημαντικό θα ήταν αυτό πανευρωπαϊκά να είχαμε μια τέτοιου είδους προσέγγιση, μια τέτοιου είδους νέα δυνατότητα δράσης γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους εγγυήσει θα διευκόλυναν λοιπόν την λειτουργία αυτών. Ένα τελικό τελευταίο ε, πράγμα το οποίο σε σχέση με συμβαστικές τροπολογίες νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια επισήμανση σχετικά είναι το θέμα της εναλλακτική χρηματοδότησης σε σχέση με τις κλασικές περιπτώσεις δανείων από τις τράπεζες για κάποια εναλλακτική δραστηριότητα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΠΑ για παράδειγμα, και στις αγορές μετοχών υπάρχουν μηχανισμοί ώστε αυτές οι αγορές να μπορούν να ενδυναμώνονται, να ε, λειτουργούν και υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να δούμε αν μπορεί να γίνει στην ε, Ευρώπη για τέτοιου είδους ε, χρηματοδοτικές δράσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια σκόπιμη δυνατότητα που θα μπορούσε να εξεταστεί προς αυτή την κατεύθυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συμβιβαστικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί νομίζω προς την σωστή κατεύθυνση στοχεύουν. Τουλάχιστον εμείς ως ομάδα αυτό πιστεύουμε και θα εγκρίνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντότμαν. Η κυρία Κλέβερ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σλοβένικα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτη αυτή για την έκθεση και την έξοχη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των συμβαστικών προτάσεων και νομίζω ότι συνέβαλαν στην ε, ενδυνάμωση της ε, εκθέσεως και ότι έχουμε πλήρη επίγνωση ενδεχομένων συνεπειών τέτοιων αλλαγών της νομοθεσίας και της λειτουργίας των διαφόρων δομών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να υποστηρίξουμε την αρχή αυτή, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασίας τους, των συμφερόντων τους. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι μέσω πλουστεύσεως των διαδικασιών θα πρέπει να μεριμνήσουμε και για την επαρκή προστασία των εργαζομένων για την ασφάλειά τους στην εργασία και για άλλα σημαντικά θέματα. Ήδη συζητήσαμε διμερώς με τον εισηγητή το ζήτημα και τα θέματα που άπτονται της συνεργασίας με τις τράπεζες και την πρόθεση διαφόρων χρηματοστατικών σχημάτων θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα κυρίως σε αυτή την εποχή. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κάτι μελη ε, ποικίλουν. Δεν υπάρχει, δεν είναι μια ομοιογενής κοινωνία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ακολουθούν και διαφορετικές πολιτικές. Όταν μιλάμε για κοινωνικές επιχειρήσεις αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Αυξάνεται το τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη είναι το 10% όλων των επιχειρήσεων. Και είναι σημαντικός εργοδότης. Θα πρέπει, λοιπόν, να μην παραλείψουμε κάποιες κάποιους νέους τρόπους να διατίθεται δημόσιοι πόροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελπίζω να βρούμε κάποιες νέες συμβιβαστικέ λύσεις με τον εισηγητή σχετικά με το θέμα. Να τονίσω εκ νέου ότι πραγματικά ήταν έξοχη η συνεργασία μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλέβερ. Ο κ. Φιλίπ Λαμπέρ είναι σκιώδης για τους Πρασίνους, αλλά δεν τον βλέπω να είναι εδώ, ούτε άλλος εκπρόσωπος των Πρασίνων. Ο κ. Καμάλ, εκ μέρους του ECR, έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την έξοχη συνεργασία μας και για την ταχύτητα με την οποία ο εισηγητή κατέληξε στι συμβαστικέ τροπολογίε είναι πρότυπο αποτελεσματικότητα. Όλοι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα. Και με τα χαρά βλέπω ότι κατανοούμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν είναι ομοιογενεί τομέα. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο το 2005, συγκλονίστηκα από τη συζήτηση ε, διότι δεν αναγνωρίζήταν ότι υπήρχε κατακαιρματισμός όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέχρι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που απασχολούν αρκετούς ανθρώπους. Είναι πολύ διαφορετικές και ένα από τα ζητήματα που είχα εγώ αντιμετωπίσει με τις δικές μου επιχειρήσεις ήταν από εκεί που ήμουν μοναδικός εμπορευόμενος να γίνω εργοδότης και να αντιμετωπίσω διάφορα θέματα που ο σκιώδης εισηγητής των σοσιαλιστών έθιξε. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι μεγαλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ανήκουν στην αλυσίδα την παγκόσμια ε, ε, φοδιασμού αν θέλετε και δεν θα πρέπει να αποκοπούμε από αυτούς. Αυτό που με ενδιαφέρει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές που είναι πολύ χαμηλά στην κοινωνία, τι φτωχότερες κοινότητες και έχουμε βλέπουμε ότι πολλοί ε, από φτωχοί με 50 λίρες, 100 λίρες με πολύ λίγα χρήματα οικοδομούν θαυμαστές εταιρείε. Υπάρχει η κυρία Μαντισάρμα, χωρισμένη, ε, δανείστηκε 10 λίρες, έφτιαξε τέσσερις σωμόσας, πιτούλες συνδικές με αυτά τα λεφτά. Ένα ορεκτικό Έβγαλε χρήματα, έφτιαχνε μετά 8 και έφτιαξε εταιρεία 16.000 σωμόζα την ημέρα. Παράγει και απασχολεί πολύ κόσμο και από την εκλογική μου περιφέρεια. Δύο παιδιά, δύο αγόρια, ε, τη δεκαετία 80 πήραν 50 λίρες για να αγοράσουν ύφασμα από την αγορά και αγόρασαν και ε, πήραν ε, τελικά την ε, ραπτομηχανή της μητέρας τους και έφτιαξαν εσώρουχα και έφτιαξαν μεγάλη εταιρεία. δείχνει ότι με ελάχιστα χρήματα μπορεί να πετύχει κανείς πολλά. Συνεργάστηκα με διάφορες οργανώσεις στη δική μου εκλογική περιφέρεια να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τόσα λίγα χρήματα σε κάποιους ανθρώπους και να τους δώσουμε ταυτόχρονα και κάποιες συμβουλές. Καλό είναι να δίνεις 50-100 λίρες ή 200 ευρώ, αλλά χρειάζονται συμβουλές αυτοί οι άνθρωποι για να οικοδομήσουν εταιρεία. Χρειάζεται και συνεργασία με τον τομέα της κατάρτισης και με διάφορα άτομα για αυτή την παροχή συμβουλών. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να δανείσουν χρήματα. Και συμφωνώ με τους σκιώδεις που είπαν ότι βλέπουμε μόνο το τραπεζικό μοντέλο. Θα πρέπει να δούμε και μεταξύ ομολόγων το δανεισμό. Το kiva.org που επιτρέπει να δανείζουμε 25 δολάρια σε επιχειρηματή στον τον κόσμο. μπορεί να βοηθήσει κάποιον στην Ουγγάντα, στην Κολομβία. 25 δολάρια δίνει ο καθένας. Αν τα θρήσει όμως από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου μπορεί να δανείζονται 1.000, 2.000, 3.000 δολάρια. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και το Kickstart, άλλη οργάνωση, που κάνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Δεν πρέπει να το πολυκουβεντιάζουμε να δούμε πώς αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να ανθίσουν τελικά. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι το εξή. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά παρεμποδίζουμε μία από τι πηγέ. Διότι συγκα... κολλησιεργούμε όσον αφορά τον κανονισμό για τα κεφάλαια κινδύνου. Απ' τη μία λέμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα χρήματα, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι που μπλοκάρουμε είναι το ευρωπαϊκό κεφάλαιο κινδύνου και όλα αυτά λόγω για λόγου φορολογικού. Είναι σημαντικό το θέμα του φόρου. Το... γίνονται μάχες για το φόρο. Ε, εντάξει, είναι σημαντικό αυτό, αλλά οι φόροι ε, δεν είναι αποκλειστικά μοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εξετάσει. Παίζουμε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αν θέλετε και τελικά το αποτέλεσμα όλου αυτού του παιχνιδιού είναι να παρεμποδίζουμε τα κεφάλαια κινδύνου που θα μπορούν να διατίθενται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να πεμπλακεί αυτή η έκθεση, να προχωρήσει να δημιουργήσουμε, να διευκολύνουμε την ε, κυκλοφορία κεφαλαίων ε, επιχειρηματικού κινδύνου στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, τελικά θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το επικοδομητικό κλίμα, για τη συνένεση, ε, για την καλή συνεργασία και για τις συμβαστικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Ούτε ο κύριος Κλιούτ είναι εδώ. Ο κύριος Μπάκαρ, θέλετε να σχολιάσετε. Ο κύριος Μπάκαρ. Πολύ σύντομα, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις τους ε, και που τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες ε, έγιναν ε, κάποια σύντομα σχόλια. Απόλυτα συμφωνώ με κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν για εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι πολλά γίνονται σε σχέση με ένα αποκλειστικό πρότυπο. Εναλλακτικέ δυνατότητε για χρηματιστήρια, μικρομεσαίε επιχειρήσει, χρηματοδότηση με δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για πιο ε, αποτελεσματικά και δίκαια τέτοια μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να εντοπίσουμε τους φραγμούς και τα προσκόμματα που παρακόλλησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν. Και στη δική μου έκθεση ένα από τα σημεία που θα ήθελα να τονίσω είναι αυτό. Ένα σημείο το οποίο είναι πραγματικά επίση σημαντικό για μένα είναι σε σχέση με τις ε, πολλές ομάδες που μπορούν να βορέσουν για τις ε, μεταφορές ε, αυτών πόρων. Να δούμε όχι μόνο τη χρηματοοικονομική πλευρά, αλλά και τη δυνατότητα με τέτοιες δράσεις να ενδυναμώσουμε τα σχέδια και τα, τον προγραμματισμό επιχειρήσεων, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για τις ρυθμίσεις του επιχειρησιακού κεφαλαίου venture capital νομίζω σε σχέση με την ε, υποβολή πρότασης ε, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα για εκείνους τους επιχειρηματίες που αναμένουν και προσδοκούν κατεπηγόντως να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να μπορέσουν να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία. Είναι επιτέλους η χρονική στιγμή να αποτροχοπεδίσουμε, να απελευθερώσουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο για να δράσουμε αποτελεσματικά. Νομίζω οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι καλύπτουν ε, πολλές τέτοιες ε, πτυχές που είναι σημαντικές και με τις συμβαστικές τροπολογίες έχουμε μια καλή έκθεση μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάκερ. Και φτάνουμε στο τέλος. Α, συγγνώμη. Πρέπει να προαναγγείλω κάτι, γιατί σχεδόν το ξέχασα. Η ψήφιση στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών θα διεξαχθεί στις 17 ή 18 Δεκεμβρίου. Και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει στην περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου. Φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Θα ξαναξεκινήσουμε το απόγευμα στις 3.15.00. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.